Αγαπητοί φίλοι, καλώ ορίσατε. Καλησπέρα. Ε, καλησπέρα, καλωσορίζω εδώ τον ε, φίλο μας τον Ματίας ε, Μπουχέρτ και τον κύριο Σμαλά. Θα μιλήσω ελληνικά. Παρακαλώ βάλτε τα ακουστικά σας. το πρώτο θέμα που έχουμε στην ατζέντα είναι η έγκριση του σχεδίου ημερησίας διαταξής. Ε, δεν υπάρχουν αντιρρήσει, οπότε το σχέδιο ημερησία εγκρίνεται. Το δεύτερο είναι η έγκριση των πρακτικών. Τα πρακτικά διαβάστηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δεν υπάρχουν αντιρρήσει, οπότε θεωρούνται εγκριθέντα. Ε, μου διέφυγε να πω στην αρχή ότι σήμερα διατίθεται ε, διερμηνία στα γαλλικά, ιταλικά, αγγλικά, ελληνικά και ισπανικά. Ε, πριν να περάσουμε στο θέμα, να μου επιτρέψετε, συνάδελφοι και φίλοι, να ε, αναφέρω σε συντομία μερικά καινούργια ε, ε, στοιχεία για την κατάσταση όπως είναι στην Παλαιστίνη. Στις αρχές του τρέχοντος μηνός η Κνέσετ ψήφισε νομοθεσία με την οποία εξουσιοτήτων Ισραηλινών Υπουργών Εσωτερικών να ανακαλεί τι άδειε μόνιμη διανομή των προσώπων που εμπλέκονται σε υποθέσει τρομοκρατία, προδοσία ή κατασκοπία. Μόνο ότι απορρίπτουν την τρομοκρατία σε όλε τι μορφέ, είναι σαφέ ότι ο νέο νόμο ενδέχεται να καταστήσει ακόμα πιο επισφαλέ από ό,τι είναι ήδη σήμερα το καθεστώ διαμονή των Παλαιστινίων στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, ενό πληθυσμού προστατευόμενου σύμφωνα με το Διεθνέ Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Σήμερα περίπου 420.000 Παλαιστίνοι στην Ανατολική Ιερουσαλήμ έχουν κάρτες μόνιμη κατοικία. Φέρουν επίση προσωρινά Ιορδανικά διαβατήρια χωρί εθνικό αναγνωριστικό αριθμό. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι πλήρης πολίτες της Ιορδανίας. Ε, για παράδειγμα, χρειάζονται άδεια εργασία στην Ιορδανία και δεν έχουν πρόσβαση σε κυβερνητικέ υπηρεσίε και κρατικέ παροχέ. Οι Παλαιστίνοι τη Ιερουσαλήμ επί τη ουσία είναι άνθρωποι δίχω ηθαγένεια, εγκλωβισμένοι σε μια κρίζα ζώνη, αφού δεν είναι πολίτε του Ισραήλ, ούτε τη Ιορδανία, ούτε τη Παλαιστίνη. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει του Παλαιστίνου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ ω ξένου μετανάστε που ζουν εκεί ω χάρη που του χορηγείται από το κράτο και όχι από το δικαίωμα και από το γεγονό ότι γεννήθηκαν εκεί. Απαιτεί από αυτού να εκπληρώνουν ορισμένο σύνολο κριτηρίων για να διατηρήσουν το καθεστώ διαμονή του και ζουν με το συνεχή φόβο ότι αυτό το καθεστώ θα ανακληθεί και θα πεταχτούν έξω από την πατρίδα του. Κάθε Παλαιστίνο που ζει εκτό των οριών τη Ιερουσαλήμ για μια ορισμένη χρονική περίοδο, είτε σε μια ξένη χώρα, είτε ακόμα στη Δυτική Όχθη, διατρέχει τον κίνδυνο να χάσει το δικαίωμα παραμονή στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Από το 1967 το Ισραήλ έχει ανακαλέσει το καθεστώ διαμονή 14.000 Παλαιστινίων, σύμφωνα με την Ισραηλινή ομάδα Πέτσλε. Ο στρατηγικό κατακαιρματισμό του Παλαιστινιακού λαού είναι η βασική μέθοδο με την οποία το Ισραήλ επιβάλλει το καθεστώ του φυλετικού διαχωρισμού ενό σύγχρονου κατά μα Απαρτχάιτ. Οι Παλαιστίνοι διαχωρίζονται και καταπιέζονται μέσω διακριτών νόμων, πολιτικών και πρακτικών. Εμεί καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυ στην εφαρμογή αυτού του νόμου για του Παλαιστίνου τη Ανατολική Ορυσαλίκη. Επίσης να αναφέρω ότι την περασμένη εβδομάδα ε, σημειώθηκε απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Παλαιστίνου Πρωθυπουργού Ραμί Χαμπτάλα στη Λωρίδα της Γάζας όταν άγνωστοι από επιτέθηκαν στην αυτοκινητοπομπή που τον μετέφερε για να παραστεί στα εγγένεια σταθμού ίδρυυση. Η επίθεση προκάλεσε ελληνικέ ζημιέ σε τρία αυτοκίνητα και σχετικά ελαφρύ τραυματισμού σε 7 άτομα τη συνοδεία του Πρωθυπουργού. Πρέπει να σα πω την ίδια και τη μέρα, απέστειλα επιστολή στον πρόεδρο τη Παλαιστίνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταδίκασα την άνδρια αυτήν πράξη και μετάφερα τη συμπαράσταση τη αντιπροσωπείας μα τόσο στον Πρωθυπουργό όσο και στου τραυματίε και ευρύτερα επαναβίωσα την ανική μα προ τον Παλαιστινιακό λαό. Την ίδια ώρα τόνισα την διαχρονική θέση ότι η ασφάλεια και η σταθερότητα στην προχή είναι κάτι παραπάνω από παρέτηση. Φίλε και φίλοι, Στη σημερινή συνεδρία θα επικεντρωθούμε στη συζήτηση για την υπηρεσία αναρρογή και έργων των ΗΕ για του Παλαιστίνου πρόσφυγε στην Αγγλική Ανατολή, την Ούρα. Όπω είπα και στην αρχή, μαζί μα έχουμε δύο αξιωματούχου. Τον Ματία Μέιλ από τη Γάζα, διευθυντή επιχειρήσεων τη Ούρα στη Γάζα, ο οποίο θα συμμετέχει στη συζήτηση μα μέσω τηλεδιάσκεψη και τον Ματία Πούρχα, τον Διευθυντή του Σούρνα στι Βρυξέλλε, ο οποίο είναι μαζί μα εδώ στην αίθουσα και του καλωσορίζουμε αναφότερου. Ε, θα ξεκινήσουμε με την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα για λόγου χρονικού περιορισμού και υλικοτεχνική υποστήριξη. Προτείνω ότι να έχουμε πρώτα μια σύντομη ενημέρωση από τον κύριο Σμέιλ από τη Γάζα και στη συνέχεια οι συνάδελφοι να του θέσουν ερωτήσει μετά την ε, λήξη της τηλεδιάσκεψης θα ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία με τον κύριο Μπούρχαρτ και θα συζητήσουμε για την οικονομική κατάσταση της Δούρα και ιδιαίτερα ενημερωθούμε για την υπουργική διάσκεψη στη Ρώμη που διεξήχθη την περασμένη εβδομάδα με θέμα διατήρηση της αξιοπρέπειας και επιμερισμός της ευθύνη, κινητοποίηση για συλλογική δράση για την Ούρα που έγινε από τη Συμπροεδρία της Ιορδανίας, της Συρίας και της Αιγύπτου. Ε, Και να δώσω αμέσως το λόγο στον ε, κύριο ε, Ματίας Νέιλ από τη Γάζα ε, να μας ενημερώσει για την κατάσταση εκεί. Κύριε Νέιλ, ακούμε ότι ενισχύουν οι εντάσεις και οι κινδύνοι κλιμάκωσης, ότι ο αποκλεισμό εξακολουθεί να δυσκολεύει υπερβολικά τη ζωή των κατοίκων του Παλαιστινιακού λαού στη Γάζα και ότι η κατάσταση γίνεται ολοένα και πια απελπιστική και βεβαίως ε, θα ακούσουμε τη δική σας ενημέρωση και βεβαίως μετά να συζητήσουμε ε, και τους τρόπους πώς μπορούμε ως αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τον Παρασυνιακό Λαό θα, ε, με την Παλαιστίνη θα, τι ενέργειες πρέπει να προβούμε για να στηρίξουμε το λαό της Παλαιστίνης που ζει στη Γάζα. Ο λόγος σε εσάς κύριε Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ελπίζω να με ακούτε καθαρά. Εκτιμάμε ιδιαίτερα την ευκαιρία αυτή που μας δίνεται να συνομιλήσετε μαζί μας ε, ε, με εμά από τη Γάζα, μαζί με τον συνάδελφο Ματία στις Βρυξέλλες. Εκτιμάμε ιδιαίτερα την πολιτική και οικονομική στήριξη από τις Βρυξέλλες το Κοινοβούλιο το Φεβρουάριο, στις αρχές του Φεβρουαρίου υιοθέτησε ένα ψήφισμα για την ΟΝΡΑ. Εκτιμάμε ιδιαίτερα πολιτικές δηλώσεις αυτού του είδους και την οικονομική υποστήριξη φυσικά. Τώρα για το πιο συγκεκριμένο θέμα τη ανθρωπιστική κατάσταση εδώ, θα ήθελα να επιθυμίσω σε όλους ότι η ΟΝΡΑ ε, έχει μεγάλη επίδραση εδώ και παρουσία στην Γάζα. Έχουμε ευθύνε για 70% του πληθυσμού 1,9 εκατομμύρια ζουν εδώ στη Λωρίδα της Γάζας 1,3 και είναι εγγεγραμμένοι στην Ούντρα Είμαστε οι κύριοι προμηθευτές ε, δημοσίων υπηρεσιών σε αυτούς τους 1,3 εκατομμύρια ανθρώπους. Ε, λειτουργούμε 275 σχολεία εδώ ε, στα οποία πηγαίνουν χιλιάδες παιδιά καθημερινά. Ε, λειτουργούμε 22 κλινικές ε, κέντρα υγείας όπως τα ονομάζουμε που είναι σαν μικρά νοσοκομεία ή μεγαλύτερα νοσοκομεία. Αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς μας εδώ. Ε, οι δημόσιες υπηρεσίες ουσιαστικά το άλλο κομμάτι που είναι σημαντικό και σχετίζεται περισσότερο με το θέμα της ανθρωπιστικής κατάστασης είναι ότι δυστυχώς, ε, όπως δείχνουν η δική μας ανάλυση, τα τελευταία δύο με τρία χρόνια τα επίπεδα φτώχειας μεταξύ των Παλαιστίνων προσφύγων έχει αυξηθεί σημαντικά κατά 15%. Αυτή τη στιγμή το 77% των Παλαιστίνων προσφύγων εδώ, δηλαδή σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι, ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Εμείς ε, αποκνόμαστε με ένα σημαντικό πρόγραμμα ανθρωπιστικό, αποτελείται από τρία ε, από τρεις συνιστώσεις. Το πρώτο είναι επισητιστική αρρωγή, παρεμβάσεις ε, σχετικές με το φαγητό. Παρέχουμε συμπληρωματικά τρόφιμα ή ουσιώδη τρόφιμα ή διατροφής σε ένα εκατομμύριο ανθρώπους κάθε τριμήνο. Το δεύτερο, η δεύτερη συνιστόσα είναι παροχή μετρητών για εργασία το ονομάζουμε πρόγραμμα δημιουργίας θέσεων εργασία. Βρισκόμαστε σε μια φθήνουσα οικονομία στη Γάζα που καταρακώνεται και μέσω από αυτό το πρόγραμμα ε, ροή μετρητών παρέχουμε ε, πάρα πολλά εκατομμύριο δολάρια. Δηλαδή πολλές χιλιάδε άνθρωποι αποφελούνται από αυτή την ευκαιρία. Για την ίδια την οικονομία αυτό είναι πολύ σημαντικό επειδή η οικονομία καταραίει αυτή τη στιγμή, αυξάνεται η ανεργία έχει φτάσει το 65% για τους νέους ανθρώπους ε, ηλικίας 15 με 29. Οποιαδήποτε λοιπόν ε, βοήθεια σε μετρητά είναι πολύ σημαντική οικονομική συμβολή. Και η τρίτη συνιστόσα της ανθρωπιστικής μας απόκρισης ε, στο πλαίσιο του προγραμματός μας είναι ένα πρόγραμμα ψυχικής κοινωτικής υγείας. Είναι σημαντικό κομμάτι αυτό όπως φαντάζεστε μετά από 10 χρόνια απομόνωσης σε μια ανοιχτή φυλακή σαν αυτή και μετά από τρεις πολέμους υπάρχουν τεράστια ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήματα. Οι δείκτες από αυτούς του, σε αυτά τα θέματα επίσης επιδεινώνονται, γίνονται όλο και πιο αρνητικοί. Όλο ένα λαμβάνουμε αναφορές από συναδέλφους μας για προσπάθειες αυτοκτονίας, ε, πριν από λίγες εβδομάδες δύο νέοι έφηβοι αποφάσισαν να τερματίσουν τις ζωές τους με διαφορά μίας ημέρας. Ήταν άσχετοι μεταξύ τους, αλλά μέσα σε δύο μέρες το ένα ήταν ένα παιδί που πηγαίνει σε ένα από τα σχολεία μας. Φαντάζεστε λοιπόν πόσο μεγάλη ήταν η αντίδραση και πόσο αυτό επηρέασε τους συμμαθητές ε, του παιδιού αυτού που την επόμενη μέρα δεν τον ε, είδαν μεταξύ τους. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική συνιστόσα αυτή. Τέλος, θα ήθελα να σας πω, επειδή είπατε να είμαστε σύντομοι για να έχουμε χρόνο για συζήτηση, ποια είναι η κατάσταση της χρηματοδότησης εδώ, ειδικότερα ε, στο ανθρωπιστικό σκέλος. Ο Ματίας, ο άλλος Ματίας της Βρυξέλλες θα μιλήσει για τη γενική κατάσταση. Σε ε, ανθρωπιστικό επίπεδο πέρυσι δαπανίσαμε 135 εκατομμύρια ε, δολάρια στη Δυτική Οχθή και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, 18 εκατομμύρια, 80 εκατομμύρια για την επισητιστική δράση όπως είπα και τα 90 εκατομμύρια από τα 135 προήλθαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τεράστια συμβολή, τεράστια εξάρτηση. Για το φετινό ετός η συμβολή τους είναι ακριβώς μηδενική. Χάσαμε δηλαδή 90 εκατομμύρια δολάρια από τη συμβολή των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι σημαίνει αυτό ότι καθώς εμείς ε, συζητάμε, εκτός αν ο έχει κάτι καλό να μας πει, δεν ε, ε, υπάρχει πλέον διασφάλιση της ανθρωπιστικής δράσης πέραν του Ιουλίου, πέραν του τέλους του Ιουνίου. Δηλαδή η διανομή τροφίμων είναι εγγυημένη μέχρι τέλη Ιουνίου. Αλλά στην παρούσα φάση δεν μπορούμε να πούμε τίποτα βέβαιο για την περίοδο μετά. Θα φαντάζεστε τι σημαίνει αυτό. Σε περίπτωση που η Ιούντρα διακόψει την διανομή φαγητού στο μισό πληθυσμό εδώ. Είναι απόλυτα σαφές ε, κατά την άποψή μου ότι από αυτή την άποψη αποτελούμε παράγοντα σταθερότητα. Αν εξαφανιστεί αυτό ο παράγοντα σταθερότητα ή μειωθεί σημαντικά, αποδυναμωθεί σημαντικά, υπάρχει περίπτωση να έχουμε ως αποτέλεσμα όχι μόνο ε, πείνα, αλλά σημαντική κοινωνική αναταραχή. Από το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών μας είπαν ότι μετά από την απόφαση του Πρόεδρου Τραμπ ε, έχουν γίνει πολύ βίες διαδηλώσεις με πολλούς τραυματισμούς ε, και πολλούς θανάτους. Φαντάζεστε λοιπόν τι θα συμβεί σε περίπτωση που διακοπεί η διανομή τροφίμων. Πιστεύω ότι υπάρχει κίνδυνος ε, να έχουμε σημαντικές αναταραχές, κοινωνικές αναταραχές και διαμαρτυρίες. Επίσης φοβόμαστε το αρκετά πιθανό ενδεχόμενο ακραίων σενάριων. Να σας ενδιαφέρει θα σας πω και κάποια παραπάνω πράγματα γι' αυτό. Τέλος, ποια είναι η λύση για κάτι τόσο δύσκολο. Νομίζω ότι η Γάζα είναι μια κατάσταση που θα μπορούσε να ανατραπεί εύκολα. Αυτό που με έχει εντυπωσιάσει τις τελευταίους ε, πέντε μήνες, ε, παρατηρώντας την κατάσταση εδώ, ε, συναντώ καθημερινά ανθρώπους με υψηλό επίπεδο παιδείας και δεξιότητες υψηλό επίπεδο και πάρα όλα τα προβλήματα εξακολουθούν να κάνουν ό,τι μπορούν καλύτερο με τις ζωές τους. Πιστεύω ότι ο κύριος παράγοντας, ο οποίος εξηγεί ότι υπάρχει ανάγκη ανθρωπιστικής δράσης και αυτός ο παράγοντας θα μπορούσε να ανατρέψει την κατάσταση ώστε να αποφύγουμε την απολύτη κατάρρευση, θα ήταν η άρση ε, του αποκλεισμού. Αν είχαμε μερικές χιλιάδες ε, ε άδειε εργασία, οι άνθρωποι θα μπορούσαν να αναζητήσουν άλλε ευκαιρίε και αυτό θα ανέστρεφε την κατάσταση, οδηγώντα σε μεγαλύτερη σταθερότητα. Ο δεύτερο παράγοντα είναι η Παλαιστινιακή Ενότητα. Σίγουρα η Παλαιστινιακή ηγεσία πρέπει να κάνει περισσότερα για να μείνει πιο ενωμένη και πιο, να γίνει πιο επικοδομητική. Υπάρχουν ευκαιρίες ε, παρότι μειώνονται. Και τρίτον, μέχρι να βρεθεί μια πολιτική λύση που θα θεωρηθεί από όλους δίκαιη, ε, και με την οποία θα συμφωνήσουν όλοι και φυσικά και οι ίδιοι οι Παλαιστίνοι. Δεν έχει νόημα να συζητάμε στη Washington πράγματα χωρίς να συμμετέχει στις συζητήσεις ο πληθυσμός ε, της Παλαιστίνης. Μέχρι να βρεθεί λοιπόν μια λύση, τα διεθνή μέσα σταθερότητας, όπως τα περιέγραψα στην αρχή και ειδικότερα η UNRWA, θα χρειαστεί να συνεχίσουν το έργο τους και επαναλαμβάνω εκτιμάμε την πολιτική και οικονομική σας στήριξη γιατί κάνει μεγάλη διαφορά στις ζωές τεράστιου αριθμού ανθρώπων εδώ. Βοηθά όμως επίσης και ε, στη διατήρηση της σταθερότητας και για τους γειτόνες, όχι μόνο για το Ισραήλ και την Αίγυπτο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για αυτή την ευκαιρία. Ευχαριστώ κύριε Σμέιλ. Νομίζω παρότι είσαστε σύντομος, είσαστε αρκετά περιεκτικός με αρκετά ε, συγκεκριμένο και υπερευτικό τρόπο δώσατε πλήρω την καταστασή. Ε, τώρα ε, απευθύνω στους συναδέλφους αν έχουν να θέσουν κάποια ερωτήματα. Ναι, ο Εντουάρ Μαρτίν. bonjour, Edouard Είμαι ο Εντουάρ Μαρτά. Σας ευχαριστώ για αυτές τις πληροφορίες. Δυστυχώς και οι πληροφορίες οι δικές μου συμπίπτουν γιατί εγώ είμαι, έχω σχέση με την Ένωση Palmed. Έχω τέτοιου πληροφορίες λοιπόν στα κτά διαστήματα και αναφέρονται οι καταστάσεις που είναι πιο σοβαρές από δραματικές αν μπορούσα να τις χαρακτηρίσω έτσι στη Γάζα. Φαντάζομαι ότι με τους συναδέλφους θα παρέμβουμε σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αντισταθμίσουμε το γεγονός ότι σταμάτησε να παρέχει οικονομική βοήθεια ε, στο επίπεδο που παρήχε μέχρι τώρα η Αμερική. Αυτό είναι κάτι το οποίο για μας είναι πρωτόγνωρο. Γνωρίζω ότι υπάρχουν κάποια δίκτυα ενώσεων που θέλουν να βοηθήσουν. Φερρυπίν, αποστείλουν φάρμακα. Το θέμα είναι ότι υπάρχει δυσκολία στην αποστολή φαρμακευτικού υλικού στη λωρίδα της Γάζα. Αυτό είναι το ένα θέμα. Δεύτερο θέμα, ερώτηση για σας. Μπορείτε να κάνετε κάτι για να διευκολύνετε αυτή την κατάσταση. Μπορείτε να είσαστε είσοδος στην οποία θα αποσταλούν στη λωρίδα της Γάζα, αν όχι, όταν η επιστημιστική βοήθεια, τουλάχιστον τα φάρμακα, η φαρμακευτική βοήθεια. Κάτι τέτοιο έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε. Yeah. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Ο συνήθω όλα θα είναι τρομακτικά και απογοητευτικά. Και πολλοί από εμά αισθάνονται τρομεροί απογοήτευση, διότι εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι ο μόνος τρόπος που μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με την Ούνρα στη Γάζα, μέσω της ε, βιντεοδιάσκεψης. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν ξέρω τι γίνεται σε επίπεδο όχι, αλλά φαίνεται έτσι όπως έχουν τα πράγματα ότι ίσως ορισμένοι σχηματίσουν την ιδέα ότι αποδέχεται αυτή την κατάσταση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει κάποια διαδικασία την οποία θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε για να μετακινηθούμε, να φτάσουμε σε εσά, επιτόπου, να δούμε μα τι γίνεται. Διότι υπάρχει αυτός ο αποκλεισμό η απομόνωση από το Ισραήλ. Ο μόνος τρόπος λοιπόν επαφή που έχουμε με εσά στη Γάζα είναι αυτή η βιντεοδιάσκεψη. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο θα ήθελα να θέσω. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται με τις διάφορες κυρώσεις οι οποίες ενδεχομένως αφορούν το Χαμάς. Νομίζω ότι θα πρέπει να εκφραστούμε με απόλυτη σαφήνεια για το θέμα αυτό ακόμη και να το συζητήσουμε με τους φίλους. Αυτοί οι οποίοι κατέχουν ένα μέρος της επικράτειας Ακούσαμε στα μέσα ενημέρωσης ότι επιτέθηκαν κάποιοι σε τρεις ε, στρατιώτες στην περιοχή σας. Βεβαίως, αν υπάρχει κάποιος ένστολος στον οποίο επιτίθενται κάπου σε μια κατεχόμενη ζώνη, είναι θέμα των μέσων ενημέρωσης. Βεβαίως αυτά είναι θέματα τα οποία ε, πέφτουν στην αντίληψή σας αν παρακολουθείτε τι γίνεται σε αυτήν την περιοχή. Διαφορετικά δεν τα μαθαίνετε. Είπατε ότι υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού που είναι εκεί στη Γάζα που έχει υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. Σας ευχαριστούμε. Εν μέρει αυτό οφείλεται σε εσά και χάρη στις δικές σας προσπάθειες γίνεται κάτι τέτοιο. Θα ήθελα να μας πείτε περισσότερα για τις προσπάθειες αλφαβητισμού που κάνετε γενικότερα και για το επίπεδο εκπαίδευσης. Διαφορετικά, θα μπορούσα να πω ότι ε, οι προσπάθειες που κάνει το Ισραήλ θα μπορούσαν να ευοδοθούν αν δεν επιδεικνύεται εσείς αντίσταση. Διότι πολλές φορές ακούμε διαφορετικές απόψεις. Βεβαίως, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε αυτό που κάνατε. Πώς μπορούμε να σας υποστηρίξουμε, πώς μπορούμε να σας υποστηρίξουμε στην προσπάθεια ενοποίησης ποιο δρόμο μπορούμε να ακολουθήσουμε για να σας βοηθήσουμε, εν πάση περιπτώσει, στο εγχείρημά σας. Ε, Φρόιντ. Ο κύριος Φρόιντ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη διότι καθυστέρησα και δεν ήμουν μόνος και ένας άλλος συνάδελφος άρχισε, αλλά εν πάση περιπτώσει μπήκαμε στην αίθουσα τη στιγμή που ε, μιλούσε ο προσκεκλημένος από τη Γάζα. Συμφωνώ με την κυρία Ουκεν βεβαίως και εγώ πρέπει να σας πω ότι Αισθάνομαι πολύ άσχημα που δεν μπορούμε να πάμε στη Γάζα. Θέλησα το προηγούμενο Σαββατοβίσματα να επισκεφθώ τη Γάζα μου απαγορεύτηκε η είσοδος όπως και στο παρελθόν όταν ε, είχα ε, κάνει διάφορες αποστολές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι κάτι το οποίο άπτεται τη γενική κατάσταση που επικρατεί στη Ρουδία τη Γάζα. Δηλαδή, επικινδυνώθηκε η κατάσταση. Δεν μιλώ για το οικονομικό σκέλος, βεβαίως, το ότι ε, μείωσαν τη συνεισφορά του στην ούνρα οι Αμερικανοί. Ξέρουμε ότι προκαλεί οικονομικό πρόβλημα, αλλά γενικότερα η κατάσταση που επικρατεί είναι η ίδια εδώ και δέκα χρόνια ή έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο το τι συμβαίνει και ε, το μόνο που μας συνδέει αυτή τη στιγμή είναι ο μικρότερος κοινός παρανομαστής για τις ενέργειές μας προς τον λαό της Παλαιστίνης. Σας εκπλήσει το ότι δεν ε, είναι παρόλα αυτά απογοητευμένοι οι άνθρωποι και ελπίζουν καλή καλύτερα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους σας για τις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας. Ρωτήθηκε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Φυσικά η συνέχιση της ε, οικονομικής υποστήριξης από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι σημαντική. Το εκτιμάμε ιδιαίτερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στείλει τη συμβολή της για το φετινό έτος και αυτό μας βοηθά. Γίνονται συζητήσεις με την ΕΚΟΝ για μια συμβολή σε ανθρωπιστικά θέματα και θα μας βοηθήσει πάρα πολύ αυτό. Ελπίζουμε να ολοκληρωθεί σύντομα η συζήτηση αυτή και να οριστούν προτεραιότητες ε, βάσει των πραγμάτων που ανέφερα εγώ να ληφθούν υπό, ε, υπόψη αυτές από την ΕΚΟΝ. Ρωτήσατε κατά πόσο η ΟΝΡΑ μπορεί να διευκολύνει την μεταφορά των απαραίτητων υλικών στη Γάζα. Ναι, έχουμε ένα προηγούμενο. Θα γνωρίζετε ότι πριν από ένα χρόνο ζήτησε, το, ζήτησαν τα Ηνωμένα Έθνη επίγοντα ε, από θέματα καυσίμου για να συνεχίσουν να τρέχουν τα νοσοκομεία. Εμείς ε, δεν λειτουργούμε νοσοκομεία, ε, αλλά λόγω της τεράστιας δυνατότητας που έχουμε στην εφοδιαστική συμφωνήσαμε να φέρουμε καύσιμα για τα νοσοκομεία και για άλλους δημοσίους οργανισμούς και για θέματα υγιεινής τους βοηθάμε λοιπόν με όποιον τρόπο μπορούμε τους εταίρους μας γιατί φυσικά τα νοσοκομεία που λειτουργούν βοηθούν τον προσφυγικό πληθυσμό της Παλαιστίνης και κάνουμε πάντα ό,τι μπορούμε για να υποστηρίξουμε όχι μόνο τους άμεσους προμηθευτές υπηρεσιών μας αλλά και τις ε, υπόλοιπες υπηρεσίες που βοηθούν τον πληθυσμό ευρύτερα. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι απαράδεκτο να μην επιτρέπεται είσοδο σε ευρωβουλευτές. Αυτό ε, λέει κάτι για τη χώρα που θεωρεί τον εαυτό τη ε, το μόνη δημοκρατία στην περιοχή δεν αφήνει του ευρωβουλευτέ να επισκεφθούν τη λωρίδα τη Γάζα. Θα το αφήσω όμω αυτό στι δικέ σα συζητήσει. Πιστεύω ότι το Ισραήλ θα πρέπει να τεθεί πρώτον ευθυνών του δημοσίω. Να σημειώσω ότι ο αποκλεισμό φυσικά λειτουργεί αμφίδρομα. Ε, ορισμένοι από εσά δεν μπορείτε να έρθετε μέσα και πολλοί κόσμοι και από εδώ θα έπρεπε να του δοθεί η ευκαιρία να βγει ενώ δεν την έχει. Όχι μόνο για τι για τις ευκαιρίες απασχόλησης όπως ανέφερα. Χθε άκουσα για έναν συνάδελφο δικό μα τη Σούνδρα, ο πρέπει να, η οποία πρέπει να υποστεί σε εγχείρηση ανοιχτή καρδιά και ο άνδρας τη δεν έλαβε άδεια να ταξιδέψει στο Αμάν για να τη παρασταθεί. Μπορώ να σας ε, πω πολλές ιστορίες που ακούμε καθημερινά για ανθρώπους που αποκλείονται από τη μία ή την άλλη πλευρά. Ρωτήσατε για το ρόλο το, του PA. Θυμάστε ότι μίλησα για προηγουμένως για διαδικασία συμφιλίωσης μεταξύ ΦΑΤΑ και ε, Χαμάσα ε, και φυσικά η Παλαιστινιακή Αρχή είναι σημαντικός παράγων σε αυτά. Εξακολουθεί να υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας ώστε η Παλαιστινιακή Αρχή να μπορέσει να αναλάβει ζωτικέ ε, κυβερνητικέ λειτουργίε εδώ. Αλλά η ευκαιρία, το πράθυρο ευκαιρία σιγά σιγά κλείνει και πιστεύω ότι οι Ευρωπαίοι ε, θα είναι σημαντικοί, σημαντικοί εταίροι. Θα πρέπει να θέσουν και την Παλαιστινιακή Αρχή Πρωτών Ευθυνών του, όχι μόνο την ΑΜΑΣ. Για παράδειγμα, οι παροχέ ηλεκτρικού ρεύματο ε, μειώνονται ε, ταχαίως και αυτό οφείλεται στην PA, στην Παλαιστινιακή Αρχή. Μπλοκάρουν κάποιες παροχές τέτοιες και αυτοί έχουν κάποια ευθύνη λοιπόν για τους ε, πολίτες εδώ και για τους πρόσφυγες ε, η Παλαιστινιακή Αρχή δεν μπορεί να παραμένει μόνο στην πολιτική διαδικασία. Θα πρέπει να βελτιώνει, να βοηθά να βελτιωθεί και η παροχή υπηρεσιών. Έχει τέτοια ευθύνη. Τέθηκε ένα ερώτημα για τη ριζοσπαστικοποίηση και τι σημαίνει αυτό. Εγώ πιστεύω ειλικρινά ότι στην παρούσα φάση η Χαμάς ε, δεν είναι η μόνη ριζοσπαστική εναλλακτική που έχουμε στη Γάζα. Έχουμε τους Ολαφιστές και τον Τάσα. Πριν δύο εβδομάδες το ISIS ε, στο Σινά, στην Αίγυπτο, δηλαδή 100 ε, χιλιόμετρα από εδώ δημοσίευσε ένα βίντεο που έδειξε, έδειχνε τέσσερις ανθρώπους, τρεις εκτελεστές ε, και δικαστές και ένα άτομο που κατηγορήθηκε για προδοσία προς την ΤΑΕΣ, προς τη Χαμάς, δίνοντας τη Χαμάς, επειδή έδωσε στη Χαμάς όπλα. Το τρομακτικό ήταν ότι και οι τέσσερις αυτοί άνθρωποι που βλέπαμε στο βίντεο στην Αίγυπτο ήταν Παλαιστίνοι. Παλαιστίνοι που έχουν εγγραφεί ως πρόσφυγες στην Ούνρα. Αν θέλετε λοιπόν να καταλάβετε τι σημαίνει η ριζοσπαστικοποίηση στην πιο ακραία μορφή, αυτή είναι. Είπα νωρίτερα ότι πιστεύω ότι το επόμενο βήμα, αν συνεχίσει να καταραίει η, ε, η, κατάσταση, θα είναι μαζική κοινωνική αναταραχή. Όταν η Χαμάς θα έχει χάσει τον έλεγχο και δεν θα μπορεί να παράσχει την ασφάλεια που παρέχει αυτή τη στιγμή, εκεί θα ανοίξει η πόρτα για πιο ακραίες εναλλακτικέ και κανείς δεν το επιθυμεί αυτό, ούτε το Ισραήλ, ούτε η Αίγυπτος. Τέλος, Κάνατε άλλε δύο ερωτήσει. Κατά πόσο έχει επιδεινωθεί η κατάσταση. Πιστεύω ναι. Μέχρι και τους πέντε μήνες που εγώ είμαι εδώ από τότε που ξεκίνησα υπήρχε κάποιος επιφυλακτικός οπτιμισμός, κάποια αισιοδοξία για την διαδικασία συμφιλίωσης. Ενώ τώρα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τους τελευταίους πέντε μήνες τίποτα δεν άλλαξε στην καθημερινή ζωή η παροχή ηλεκτρισμού ε, είναι καλύτερη, δεν είναι καλύτερη, οι, οι δεν είναι ευκολότερες, πολλοί δείκτες έχουν επιδεινωθεί, η κατάσταση γενικώ ε, έχει επιδεινωθεί, έχουμε μεγαλύτερη ενεργεία, μεγαλύτερο ποσοστό αυτοκτονιών, όλα αυτά δημιουργούν ανησυχίες. Μετά τέθηκε το ερώτημα του πού υπάρχει ελπίδα. Δεν μπορώ παρά να επαναλάβω ότι ο λαός της Γάζα ε, επιδεικνύει τεράστια αντοχή Φαντάζομαι ότι γνωρίζετε τι σημαίνει αντοχή θεωρητικά, αλλά πρέπει να το δείτε ερχόμενοι εδώ στη Γάζα να σα επιτραπεί η είσοδο. διότι η εμπειρία αυτών των ανθρώπων που δεν έχουν ακόμα καταρρεύσει είναι εντυπωσιακή. Αλλά υπάρχει κίνδυνο υψηλό να επιδεινωθεί η κατάσταση να καταρρεύσει. Εγώ ελπίζω ότι από Ισραηλινή πλευρά, από αμερικανική πλευρά και από πλευράς διεθνού κοινότητα αλλά και από πλευρά Παλαιστινιακή αρχή, οι άνθρωποι θα λογικευτούν και θα κάνουν επιτέλους κάτι το οποίο θα διευκολύνει να αρθεί ο αποκλεισμό. Υπάρχουν όλα τα μέτρα, όλες οι συνθήκες για να αναζωογονηθεί η οικονομία συμπεριλαμβανομένης της απλής, για παράδειγμα, επέκτασης της αλλιευτικής ζώνης. Πολλοί άνθρωποι είναι αλληλείς. Αν επεκτείνουμε την αλλιευτική ζώνη κατά 2 με 3 χιλιόμετρα ή 4 χιλιόμετρα, αυτό θα κάνει μεγάλη διαφορά με την άσκηση πολιτική πίεση σε όσου έχουν πολιτική ευθύνη από αμφότερε πλευρέ για να μπορέσει να βελτιωθεί κάπω η κατάσταση. Ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία. Ε, ε, ευχαριστώ κύριε Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι πολύ σύντομα γιατί πρέπει να συνεχίσουμε. Εγώ προσπάθησα να είμαι πολύ σύντομος προηγουμένως. Μιλήσατε πολύ για το θέμα της ηλεκτροδότησης και για τον ρόλο τον οποίο παίξατε εσείς για τη μεταφορά καυσίμων για την ηλεκτροδότηση των νοσοκομείων. Έχουμε να κάνουμε με πολλά εκατομμύρια δολάρια. Το δίκτυο ιατρών στην Γάζα ε, θέλουν να κάνουν ένα, ε, μια ηλιακή εγκατάσταση ε, για την παραγωγή ρεύματο δεν έχουν χρήματα, αλλά λείπει και, το, λείπει και ο εξοπλισμό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορείτε να κάνετε κάτι. Επίσης, όσον αφορά τη ριζοστικοποίηση, είπατε ότι δεν θέλει κάτι το Ισραήλ. Εγώ νομίζω ότι αντιθέτως παίζει το παιχνίδι του το Ισραήλ. Και η Νταέσο όσο περισσότερα φαινόμενα ριζιαστικοποίησης ε, εμφανίζονται, τόσο περισσότερο παίζει το παιχνίδι και... Κύριε ε, σε σχέση με τον ηλεκτρισμό, επειδή άκουσα, υπάρχει ε, κάποιες σκέψεις για να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά για παροχή ηλεκτρισμού στα νοσοκομεία. Ε, για, για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με την έλλειψη ηλεκτροδότηση και καύσιμα. βεβαίω, αντιλαμβάνομαι ίσω, Έντουαρ να είναι και αυτό μια πρόταση που μπορούμε να σπρώξουμε για να γίνει η χρηματοδότηση για τέτοια αργά από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω έγινε με τη μονάδα αφαλάτωση. Γιατί όντω ε, στα νοσοκομεία πήγε η παροχή ηλεκτρισμού. Ε, Απλώ ήθελα να συμπληρώσω εγώ αυτό που είπε ο Έντουαρ. Ο λόγο εσά, κύριε Σμέχλ. Um, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα ότι η ηλιακή ενέργεια και οτιδήποτε μειώσει την εξάρτηση από τις παραδοσιακές μορφές ενέργειας θα βοηθήσει τη Γάζα. Όπως σας είπα, εμάς, ο κύριος στόχος μας δεν είναι να βοηθήσουμε κι άλλες ενώσεις με τα σχέδιά του, διότι πραγματικά έχουμε ε, εμείς ε, τα δικά μας προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, αν γίνει κάτι τέτοιο, μπορούμε να διευκολύνουμε τέτοιου είδους ε, σχέδια. Είτε αφορούν την ηλιακή ενέργεια, είτε αφαλάτωση, εν πάση περιπτώσει. Όταν ε, έρθει η ώρα της εφαρμογής, μπορούμε να βοηθήσουμε. Όσον αφορά το ενδιαφέρον του Ισραήλ. Ειλικρινά πιστεύω ότι η κοινωνία ε, στο Ισραήλ είναι χωρισμένη για τέτοιου Ε, Και ίσως θα το βρείτε και θέματα ασφαλείας παράξενο. Δεν θέλουν να υπάρξει καμία έκρηξη στην περιοχή της Γάζας, διότι θα υπάρχουν ε, τρομερές επιπτώσεις. Για δικούς τους λοιπόν εγωιστικούς λόγους δεν θέλουν πολύ στο Ισραήλ να αλλάξει τίποτα. Θέλουν ε, να υπάρξει σταθερότητα στη Γάζα. Γι' αυτό πολλές φορές εμφανίζονται και ως φίλοι των Παλαιστινίων για πραγματιστικούς λόγους. Πιστεύω λοιπόν ότι μπορούμε ε, για κάποια θέματα να συζητήσουμε μαζί τους για να μην ε, κραγεί η κατάσταση και εκτροχιαστεί περισσότερο. Νομίζω λοιπόν εν περιλήψει ότι δεν είναι μόνο θέμα Ισραηλινής πλευράς το ότι δεν μπορούμε να έχουμε συζητήσεις για την βελτίωση των συνθήκων ζωής στη Γάζα. Νομίζω ότι και η Ισραηλινοί αλλά και οι Παλαιστίνοι πρέπει να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε προσπάθεια βελτίωσης γίνει. ε, θέλω να παραλάβω αυτά που αναφέρετε στο κλείσιμο σας ότι Όντω η κατάσταση στη Γάζα μπορεί να ανατραπεί εύκολα. Και συμφωνούμε ότι το πρώτο είναι ένα ο αποκλεισμό. Και είναι εδώ που εργαζόμαστε βεβαίω με τι δυνάμει που έχουμε και εδώ στο Κοινοβούλιο για να, κυρίως, να ασκήσουμε την επιρροή μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να δουλέψει μαζί με τη διεθνή κοινότητα για αρθεί ο αποκλεισμό. Το δεύτερο, η Παλαιστινιακή Ενότητα, και να σα πω κύριε Μέρη, σε όλε τι συναντήσει που έχουμε και εδώ και στην ε, Ραμάλα και στη Δυτική με αξιωματούχους ε, της ε, Παλαιστινιακής Αρχής με εκπροσώπους από πολιτικά κινήματα είναι κάτι που τονίζομαι πάντοτε. Για μας είναι πολύ σημαντικό, κάτι που το συζητήσαμε εκτεταμένα και στην περσινή μας επίσκεψη, θεωρούμε την Παλαιστινιακή Ενότητα πολύ αναγκαία στη σημερινή κατάσταση για να αρθούν τα προβλήματα και να ε, επιτευχθεί ο στόχος που θέτουν οι Παλαιστίνοι για ε, να έχουν Παλαιστινιακό κράτος. Ε, το τρίτο είναι αυτό που είπατε με την ούρα, είναι κάτι που θα συζητήσουμε στη συνέχεια με τον κύριο Μπούρχαρτ ε, και πώς εμείς ως Κοινοβούλιο συμβάλλουμε πέραν από το ψήφισμα που παραφέρεται στην αρχή που ήταν ένα σημαντικό βήμα και να πω ότι είχε την έγκριση της συντριπτικής πλειοψηφία του Κοινοβουλίου από, από τις περισσότερες τουλάχιστον πολιτικές ομάδες και από την πλειοψηφία των μελών και εύχομαι και ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να σας συναντήσουμε εκεί στη Γάζα. Η αλήθεια είναι ότι με τις επισκέψεις μας στην Παλαιστίνη ε, έχουμε τη δυνατότητα και βλέπουμε ε, ε, τη δουλειά που κάνει η ΟΥΡΑ. Επισκεφτήκαμε πολλές φορές προσφυγικούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη. Ξέρουμε ότι χωρίς την παρουσία και τη συμβολή της ΟΥΡΑ οι συνθήκε θα είναι δραματικές για τους ανθρώπους Ευχόμαστε και ελπίζομαι, είπαν και άλλοι συναδέλφοι, να σα πω ότι εγώ τουλάχιστον τα τελευταία ε, τέσσερα χρόνια μετά το 2014 είναι πέντε φορέ που αιτήθηκα ε, την ε, άδεια για να πάω στη Γάζα, όπω και άλλοι συναδέλφοι. Δεν δυστυχώ υπάρχει αυτό ο αποκλεισμό και για εμά τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, πράγμα που θεωρούμε απαράδεκτο και το καταγγείλαμε πάρα πολλέ φορέ και δημόσια. Σας ευχαριστώ και πάλι κύριε Σμέιλ και ε, θέλω να ελπίζω να εκφράζω όλα τα μέλη της ε, αντιπροσωπείας ότι είμαστε δίπλα σας ε, στο δύσκολο έργο που έχετε εκεί για να αντιμετωπίσετε πραγματικά μια μεγάλη ανθρωπιστική κρίση. Ευχαριστούμε και πάλι κύριε Σμέιλ. Ε, τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, θα συζητήσουμε με τον κύριο Ματία Μπούρχαρτ, τον Διευθυντή τη Υπηρεσία Αρρωγή και έργο των ΗΕ για του Παλαιστινίου πρόσφυγε στην Εγγύη Ανατολή, την Ούρβρα. Ε, Στι 15 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η Υπουργική Διάσκεψη στη Ρώμη. Ε, ήταν η διάσκεψη για τη διατήρηση τη αξιοπρέπεια και επιμερισμό τη ευθύνη, κινητοποίηση για συλλογική δράση για την Ούρβρα από τη, υπό τη συμπροεδρία τη Ιορδανία, τη Σουηδία και τη Αιγύπτου. Η Ούνδρα σήμερα αντιμετωπίζει την πιο δύσκολη οικονομική κατάσταση από τότε που ιδρύθηκε το 1949 και γνωρίζουμε ότι η επιδίωξη τη της Ρώμης ήταν η διεθνής κινητοποίηση προκειμένου να βοηθηθεί η Ούνρα στη χρηματοδότηση του υπηρεσιακού προπολογισμού τη. Χωρί αυτή τη χρηματοδότηση δεν θα είναι πλέον σε θέση να παρέχει υπηρεσίε δοτική σημασία σε εκατομμύρια Παλαιστίνους πρόσφυγες Και νομίζω ακούσαμε προηγουμένω τον κύριο Σμίλ ότι ε, η, ε, η επισυστοστικό πρόγραμμα φτάνει μέχρι τον Ιούνιο για την Γάζα και αφορά 1,3 εκατομμύρια ανθρώπου εκεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταστεί ο μεγαλύτερο και πλέον αξιόπιστο δωρητή τη Ούνδρα μετά την απόφαση των ΙΠΑ να περικόψουν πάνω από το ίμιση τη προβλεπόμενη χρηματοδότηση. Πρέπει να σα αναφέρω, κύριο Πούρχατ, ότι και να το γνωρίζουν και τα μέλη, ότι τελευταίε μέρε η αντιπροσωπεία μα ετοίμασε ε, το γραφείο δηλαδή τη αντιπροσωπεία, εγώ μαζί με τι δύο αντιπρόεδρου, την ε, Μάρκαρετ και την Μαρίδα, ε, επιστολή που θα αποστείλουμε στην Αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την είπα την εκπρόσωπο την κυρία Μονκερίνη και στον Επίτροπο για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινωνία τον κύριο Ιωάννη Χάν, ζητώντα του να αναλάβουν επιπλέον δεσμεύσει προ την ούρα στην παρούσα κατάσταση. Για μα είναι θέμα αρχή. Η διακοπή τη χρονοδότηση τη ούρα αποτελεί τίμα των προσπαθειών αποσταθεροποίηση που έχουν στόχο να εξαλείψουν κατά την άποψή μα και την προοπτική τη του κρατών. Δηλαδή, που στιγμή που νομίζω ακούσαμε τον κύριο Σμίλ, τι συνέπειε θα έχει εάν ε, σταματήσουν τα προγράμματα σύνορα στην Γάζα. Ε, και γι' αυτό είχαμε ζητήσει την επιπρόσθετη, ζητούμε την επιπρόσθετη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτό από τη δεσμεύση τη Επιτροπή, να επισπεύσει την προγραμματισμένη συνεισφορά για το 2018 και έχοντα κατά νου ότι η υπηρεσία έχει υποσχεθεί να ξεκινήσει η ενδελεχή διαδικασία εσωτερική μεταρρύθμιση, βεβαίω κάτι που μπορείτε να μα ενημερώσετε. Και γι' αυτόν ο λόγο σε εσά, κύριε Πούτχαρτ, ε, έχετε 10 λεπτά για να μας ενημερώσετε και για την συνάντηση, τη διάσκεψη της Ρώμης. Thank you so much. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρο, κύριε Αντιπρόεδρο, σας ευχαριστούμε που με καλέσατε. Θα ήθελα, αν με ακούν και συνάδελφοι από τη Γάζα, να τους ευχηθώ ότι καλύτερο. Θα σας δείξω ένα βίντεο δύο λεπτών από την συνάντηση στη Ρώμα. Στη Ρώμη, στην οποία είχαμε 300 προσκεκλημένους. Δύο λεπτά λοιπόν θα δείτε το βίντεο της Ρώμης. الوزراء سعادة الأمين العام المندوبون الموقرون اسمي أحمد وأنا أمين سر برلمانات الأنور والمدرسية وقد تم انتخابي من قبل أكثر من نصف مليون طالب وطالبة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 إن كرامتنا لا تقدر بثمن Thank you. Uh, it Ευχαριστούμε. Όπως προαναφέρθηκε, πρέπει να δούμε τι ποια είναι τα διακυβεύματα σήμερα. Προσπαθεί να σας το δείξει το σχολείο αυτό. Τι Ποιο είναι το διακύβευμα λοιπόν με την υποχρηματοδότηση. Κυρίως το πάνω από μισό εκατομμύριο παιδιά τα οποία πηγαίνουν καθημερινά στα 75.000 σχολεία που έχουμε. Είναι η ιατρική περίθαλψη την οποία παρέχουμε. Είναι το ρευστό που δίδεται στους Παλαιστινίους, 1 εκατομμύριο επτά η επιστημιστική δίστη Οποιαδήποτε βοήθεια, αρρωγή μπορούμε να παράσχουμε στην ε, δυτική, στην ε, λωρίδα της Γάδας, στο Λίβανο, σε άλλες χώρες. Οι απειλές, τα θέματα ασφάλειας, οι απειλές από την ε, ριζοστικο... ριζοσπαστικοποίηση. Όλα αυτά λοιπόν είναι τα διακυβέρματα, όλα αυτά τι τίθενται κινδύνο. Θα πρέπει επίσης να υπενθυμίσω κάποια θέματα που αφορούν τα γεγονότα. Στις 17 Δεκεμβρίου πέρσι, πολύ πρόσφατα, υπογράσαμε ένα, μια συμφωνία πλαίσιο με τη ΣΥΠΑ, στην οποία αναγνώρισαν ρητά ότι είναι σημαντικό να μας παρέχουν ε, κονδύλια επαρκή για να φέρουμε σε πέρα στην εργασία μας. Και ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένοι για τον τρόπο με τον οποίο ενεργούμε. Και μας είπαν ότι θα λάβουμε το ίδιο ποσό το οποίο είχαμε λάβει και πέρσι. Περίπου δηλαδή 360 εκατομμύρια, εκατομμύρια δολάρια. Στις 16 Δεκεμβρίου λοιπόν μας ανακοινώθηκε ότι θα πάρουμε μόνο 60 εκατομμύρια και η επόμενη δόση 65 είναι υπομελέτη. Δεν έχουμε ακούσει να λέγεται τίποτα. Στις 17 Ιανουαρίου ο ο Γενικός Υπεύθυνος έκανε μια δραματική έκκληση στην όλους και στις 21 Ιανουαρίου είχαμε μια έκτακτη συνάντηση με τους δωρητές στο ΑΜΑΝ και ζητήσαμε να οργανωθεί μία διεθνής διάσκεψη ώστε να κινητοποιηθούν για την ούνρα οικονομικά όλοι οι υπεύθυνοι. Αυτό είναι κάτι το οποίο καταλαβαίνετε ότι επηρεάζει πολύ την όνρα. Ο επικεφαλής μας επισκέφθηκε το Ριά, το Όσλο, το Χόλμη, το Μονάχο, το Λονδίνο, το Ντουμπάι, τη Γενέβη, τη Ρώμη, το Τόκιο και άλλες πόλες πρόσφατα συνάντησε 21 υπουργούς, την ανώτατη αξιωματούχο κυρία Μογκερίνη, τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας Μακρόν και βεβαίως τελευταία, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό βεβαίως, τον Πάπα. Όλα αυτά έγιναν ενώ συγχρόνως η ΦΑΟ δέκτηκε να ε, οργανώσει για μας αυτή την ε, συνάντηση που έγινε στη Ρώμη για τη διατήρηση αξιοπρέπειας και τον εμπερισμό των ευθυνών που οργανώθηκε τις 15 Μαρτίου στη Ρώμη. Ποτέ στο παρελθόν δεν είχε υπάρξει μία τέτοια μεγάλη έκφραση πολιτικής υποστήριξης και δημοσιότητας που δόθηκε όσο για αυτή την ε, διάσκεψη που είχαμε στη Ρώμη. Είχαμε 77 ε, αντιπροσωπείες, ε, είχαμε την ε, συμπροεδρία της Ιορδανίας, της Σουηδίας, της Αιγύπτου. Είχαμε την παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, την κυρία Μογκερίνη, ο Πρωθυπουργό της Παλαιστίνης, ο κ. Σαπτάλα, ήταν εκεί, ο Γενικός Γραμματέας της Οργάνωσης Ισλαμικών Κρατών, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας της Αραβικής Ένωσης καθώς και περίπου 47 υπουργοί ε, παρέστησαν και όλοι έκαναν έκκληση και είπαν ότι πραγματικά ανησυχούν για την κατάσταση στην Παλαιστίνη και είπαν πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η Ούνρα για την ε, επιβίωση των Παλαιστινίων. Εκφράστηκαν επίσης ανησυχίες για αυτή την άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση και έγιναν πολλές αναγγελίες όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Έγιναν δεσμεύσεις για την παροχή περαιτέρω κονδυλίων. Πρέπει να πω ότι μέχρι τώρα έχουμε νέες συνεισφορές της τάξης των 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Μεταξύ άλλων, εδώ συμμετείχαν χώρες όπως η Τουρκία, ο Καναδάς, το Κατάρ, η Ινδία, η Ελβετία, η Γαλλία, η Νορβηγία, η Κορέα, το Μεξικό και η Εστονία. Πολλές αυτές είπαν ότι όντως ε, θα, πρέπει, θα αποστείλουν τα χρήματα, αλλά πρέπει εμείς να κάνουμε διπλό έλεγχο για να δούμε ποιος τα έχει αποστείλει. Και βεβαίως πολλές χώρες εξέφρασε την πρόθεσή τους να, δώσουν, να αποστείλουν περισσότερα κονδύλια και ελπίζουμε ότι σύντομα θα αναγγείλουν κάτι τέτοιο. Πρέπει να πω ότι αυτό ήταν ε, κάτι το πολύ σημαντικό, ήταν το πολύ σημαντικό πρώτο βήμα, αλλά όπως χρειά, ξέρετε χρειαζόμαστε 446 ε, ε, εκατομμύρια δολάρια, έχουμε μόνο 100 μέχρι τώρα και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε με διάφορες δραστηριότητες και σχέδια να μειώσουμε το έλλειμμα αυτό που έχουμε. Στις 15 Μαΐου ε, θα έχουμε συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για να δούμε ποια είναι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί και τον Ιούνιο με τη Συμβουλευτική Επιτροπή θα δούμε ποια πορεία θα ακολουθήσουμε. Τελικά, οι οικονομικές δεσμεύσει που ανελήφθηκαν ελπίζουμε ότι θα ξεπεράσουν αυτά τα 100 εκατομμύρια και ελπίζουμε ότι θα έχουμε αρκετά κονδύλια ε, ως το καλοκαίρι για να κλείσει η σχολική χρονιά. Μετά όμως το τι θα γίνει είναι ερωτηματικό. Δυστυχώς για σας Γάζα δεν έχω καλά νέα να μεταφέρω. Ελπίζω όμως ότι μπορώ να σας πω ότι υπήρξαν πάρα πολλές καλές προθέσεις, έγινε μεγάλη κινητοποίηση εκ μέρους αυτών των 77 χωρών που συμμετείχαν στην ε, διάσκεψη της Ρώμης και τώρα θα πρέπει να παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγες τι κάνουν για να μπορέσουν αυτά τα λόγια και τις δεσμεύσεις να τις κάνουν έργα. Και ελπίζουμε ότι και η ανθρωπιστική βοήθεια θα φτάσει στη Γάζα, διότι όλοι αναγνώρισαν, όπως και εσείς είπατε, πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό για την ε, ασφάλεια και όχι μόνο για την Γάζα αλλά και για όλες τις γειτονικές χώρες ε, στην περιοχή. Για μην αναφερθώ ιδιαίτερα μόνο στο Λίβανο, στην Ιορδανία και στη Λόρια της Γάζα. Μας απασχολεί όλους ιδιαίτερο στο όλο θέμα. Και πριν να ολοκληρώσω θα ήθελα να ευχαριστήσω όπως και ο Ματίας από τη Γάζα την Ευρωπαϊκή ε, Ένωση για την ε, βοήθεια που μας παρέχει. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ψήφισμα της 8 Δευτέρου και για την υποστήριξή του γενικότερα. Πρέπει να σας πω ότι σε όλες αυτές τις προσπάθειες που γίνονται σε διπλωματικό μεταξύ άλλων επίπεδο τις τελευταίες εβδομάδες, βλέπουμε και ενημερώνουμε και εσείς μπορείτε να ενημερώσετε τις κυβερνήσεις της χώρας σας για την μεγάλη κινητοποίηση και την αλληλεγγύη. Ξέρουμε ότι ε, μας έχει δώσει ως προκαταβολή ήδη ένα μεγάλο ποσό η Ευρωπαϊκή Ένωση φέτος. Αυτό είναι εξίσου σημαντικό. Και έτσι το ότι τα επόμενα τρία χρόνια ε, είναι εγγυημένα τα ποσά τα οποία προκαταβάλλονται και καταβάλλονται γενικότερα ε, στην ε, ούνρα είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό και βεβαίως είναι πάρα πολύ γενναιόδορη η συνεισφορά τους. Η επιστολή σας λοιπόν κύριε Πρόεδρε στον Επίτροπο Χάνα και στην κυρία Μογκερίνη είναι ιδιαίτερα επίκαιρη και σας ευχαριστούμε διότι έτσι μπορούν να δουν με ποιο τρόπο μπορούν να μας βοηθήσουν σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που είμαστε. Ε, ο λόγος τώρα στους συναδέλφους. Ευχαριστούμε για αυτές τις πληροφορίες. Όπως είπε ο Πρόεδρος, μπορείτε να υπολογίσετε στη βοήθειά μας και θα προσπαθήσουμε σε όλα τα επίπεδα να συλλέξουμε τα κονδύλια αυτά το συντομότερο δυνατόν, διότι όπως λέτε είναι πήγοντα τα θέματα. Εγώ ήθελα να σας κάνω μια άλλη ερώτηση, ήθελα να την κάνω στους συναδέλφους ε, στη Γάζα, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Ε, όπως ανέφεραν και οι συνάδελφοί σας, ε, είναι δύσκολο να συσταθεί το ιατρικό σώμα στη Γάζα. Υπάρχουν γιατροί, αλλά χρειάζονται ειδίκευση ειδικότερα σε ε, χειρουργία καρδιάς, ε, καρκίνο κτλ. Και όπως είπαμε ε, υπάρχουν, αυτό οφείλεται στις δυσκολίες εξόδου από τη Γάζα, αλλά ακόμη και αν καταφέρουν κάποιοι γιατροί να φύγουν από τη Γάζα και να έρθουν στην Ευρώπη για εκπαίδευση, αντιμετωπίζουν μια άλλη δυσκολία, την βίζα, τη θεώρηση. Και η δική μου χώρα, η Γαλλία, δυστυχώς δεν αποτελεί εξαίρεση, τους δίνει τουριστικές θεωρήσεις το να εκπαιδεύεται λοιπόν ένα ε, γιατρό σε χειρουργία καρδιά ε, είναι κάτι πολύ περίπλοκο. Έχουμε ρωτήσει διάφορε κυβερνήσει. Φαντάζομαι ότι και εσεί θα το γνώριζετε το, το πρόβλημα αυτό. Διότι τίθε το πρόβλημα της τροφοδοσίας φυσικά, του ηλεκτρικού ρεύματο, αλλά και το πρόβλημα της κατάρτισης του ιατρικού προσωπικού. Η UNRWA λοιπόν παίζει κάποιο ρόλο, μπορεί να διευκολύνει τις εξόδους στην υποδοχή στις ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία και άλλες που υποδέχονται αυτούς τους εκπαιδευόμενους ιατρούς, ε, αλλά τους δέχονται μόνο για σύντομες ε, περιόδους ε, που επιτρέπουν οι τουριστικές θεωρήσεις. Εδώ εμείς ζητάμε τη δική σας βοήθεια. Να πείτε εσείς, να, για ανθρωπιστικούς λόγους επίσης έρχονται αυτοί οι γιατροί στην Ευρώπη από τη Γάζα για να μπορέσουν να εκπαιδευτούν και να είναι σε θέση να παρασχούν ιατρικές υπηρεσίες στους κατοίκους της Γάζας. Έχετε τέτοια αρμοδιότητα Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ ε, για την παρουσίασή σας και για τις ε, ακούραστες προσπάθειές σας ε, να συμμετέχετε σε αυτές τις διασκέψεις, να συλλέγετε τα χρήματα. Ευχαριστώ και τους συνοδέλφους που συμφώνησαν για αυτό το ψήφισμα όπου ε, και τα έξι κόμματα αποφασίσαμε να δείξουμε ότι δεν πολιτικοποιούμε την ανθρωπιστική βοήθεια. Όπως το είπατε και εσείς ε, και το καταστήσατε σαφές το πώς ε, βλέπατε τα πράγματα το Δεκέμβριο, αλλά φυσικά τα πράγματα εξελίσσονται διαφορετικά από ό,τι προβλέψαμε, όπως γνωρίζουμε. Αυτό που θα με ενδιαφέρε έγινε μια συνάντηση στο Μόναχο, στην διάσκεψη ασφαλείας του Μονάχου στη Γερμανία ε, την πρώτη εβδομάδα. Υπάρχει κάτι από τη Γερμανία, όπως γνωρίζετε εσείς, το έχουν συμπεριλάβει στο έγγραφο του συνασπισμού ε, το, να υποστηρίξουν την ούνδα Τώρα πέραν αυτού έχουμε τη διάσκεψη στο Skype και τα λοιπά μπορούμε να κάνουμε τέτοιε διασκέψει με τα σχολεία, αφού δεν μπορούμε να πάμε δηλαδή, δεν παίρνουμε άδεια για να πάμε στη Γάζα, αφού δεν μπορούμε να επισκεφθούμε τα σχολεία που υποστηρίζουμε, δεν μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με τους μαθητές. Μέσω αυτή τη επιτροπή ή κάποιες άλλες ε, να απαντήσουμε ερωτήσεις ε, των μαθητών, αφού δεν μπορούμε να επισκεφθούμε τα σχολεία. Να ρωτήσουμε λοιπόν το μαθητικό σώμα, να μας πούν όλοι αυτοί οι αφοσιωμένοι μαθητές που θα μπορούσαν να μας έτσι να μας κάνουν ερωτήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πιστεύω θα τους άρεσε αυτή η ιδέα, να έρθουμε σε επαφή με αυτούς τους μαθητές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Η Μάρκαρτ. <coughs> Λοιπόν, εγώ αναρωτιόμουν, επειδή θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο το ότι δεν μπορούμε να πάμε Παλιότερα πηγαίναμε τακτικά στη Γάζα. Πολλά χρόνια κάνω εγώ αυτή τη δουλειά και έχω πάει στη Γάζα πολλές φορές και ξαφνικά δεν με επιτρέπεται είσοδος. Και εγώ δεν ξέρω τι να κάνω. Και μα... Έχω την αίσθηση ότι κανείς δεν κάνει τίποτα. Είναι απαράδεκτο να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δύο μέρε χρειάζεται για να πάρει κανεί από τη Ράφα. διότι η κατάσταση ασφαλείας ε, στην Αίγυπτο φυσικά τώρα είναι καλύτερη από ό,τι ήταν τελευταία φορά που συζητήσαμε. Παρότι λοιπόν το θεωρώ απολύτως απαράδεκτο το ότι έχουμε τέτοια προβλήματα, και έχουμε και την έκκληση από τη Γάζα ότι πρέπει να κάνουμε κάτι για να διευκολυνθεί η συμφιλίωση, η επανένωση. Είναι κάτι απολύτως αναγκαία όλο αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς βοηθά αυτή τη διαδικασία. Τη μία βοηθά την άλλη όχι. Εγώ σοκαρίστηκα την περασμένη εβδομάδα. Είδα ξαφνικά ένα tweet από κάποιον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο οποίος επιτίθετο στην Αναγκόμες. Η Κομισιόν τώρα δηλαδή παίρνει θέση υπέρ του δεξιού Ισραήλ και μας κατηγορεί για μια διάσκεψη που κάναμε από απόσταση. Τι γίνεται. Αυτό πρέπει να μπει και στα πρακτικά. Και το άτομο που το έκανε αυτό πρέπει να πουληθεί άμεσα ε, από τον Τίμερμαντς. Εγώ πήγα και την έψαξα στο Google και την πληρώνει ο Τίμερμαντς. Γιατί το δεχόμαστε αυτό. Θα πρέπει να δείξουμε μεγαλύτερη σκληρότητα. Παλιότερα είχαμε μεγαλύτερη υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία εξωτερική Δράσης και ξαφνικά δεν έχω την αίσθηση ότι συμβαίνει το ίδιο. Ναι, ωραία είναι τα χρήματα βέβαια. Παρατήρησα ότι δεν αναφερθεί και η Δανία γιατί εμείς ήμασταν αρκετά ψηλά στο κατάλογο αυτό. Τι κάνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής δράση. και όταν ξαφνικά κάποιο, κάποιο ε, υπάλληλο τους ε, επιτίθεται σε ένα μέλο μας εδώ και αυτό ε, αποστέλλεται και με tweet ε, στην, από την πρεσβεία της Ευρωπαϊκή Ένωση στο Τελαβίβ. Πώς είναι δυνατόν. Ευχαριστώ, έχω μιλήσει ήδη με την Αναγκόμες είπε ότι αυτή θα διαμαρτυρηθεί στον Ταγιάννη και στον πρόεδρο, στον πρόεδρο της Κομισιόν επίσης. Έχει στείλει επιστολή για, αυτό τον υπάλληλο, για αυτή την υπάλληλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Μπουχάρτ, έχετε το λόγο. Να κάνω ένα σχόλιο μόνο για τα όσα είπε ο συνάδελφος ο κ. Λίτς. Καλή ιδέα είναι πράγματι να το συζητήσουμε εδώ. Δεν μπορούμε να πάμε να επισκεφθούμε τη Γάζα, αλλά θα μπορούσαμε να φέρουμε κάποιε εικόνε από τη Γάζα εδώ, μέσω τηλεδιάσκεψη. Είναι ο μόνο τρόπο. Καλή ιδέα, ναι, πράγματι. Να κάνουμε αυτή την τηλεδιάσκεψη, με τα, τη βιντεοδιάσκεψη με τα σχολεία. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Δεν είμαστε πλέον συνδεδεμένοι, φαντάζομαι, με του συναδέλφου από τη Γάζα. Δεν θα είναι εύκολο για μένα να απαντήσω κυρίως στις ερωτήσει που του αφορούν, δεδομένου ότι αυτοί γνωρίζουν το θέμα πολύ καλύτερα. Αλλά από την εμπειρία μου μπορώ να πω ότι όλοι πραγματικά σεβόμαστε αυτή τη σκελεσίδα. Η Ούνρα δεν έχει την δυνατότητα, διότι έχουμε τόσο πολύ περιορισμένο προσωπικό, αλλά και η εντολή που μας έχει δοθεί είναι τέτοια που δεν μπορούμε να αρχίσουμε διαπραγματεύσεις με κάθε χώρα χωριστά για θέματα ε, ταξιδιωτικά θεωρήσεων. Δεν συμμετέχουμε σε τέτοιου είδους θέματα, δηλαδή να ζητήσουμε θεωρήσεις Schengen. Ίσως δεν σας κατάλαβα καλά. Νόμιζα ότι κάτι τέτοιο θέλατε να ζητήσουμε. Όχι, όχι. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση. Ίσως να στείλουμε μία επιστολή ευαισθητοποίησης, αν θέλετε, στα 28 κράτη-μέλη θα θέλαμε να πούμε ότι τα άτομα τα οποία έρχονται στην Ευρώπη έρχονται για κατάρτιση και μετά γυρίζουν πίσω στη Γάζα. Απλώς να ευαισθητοποιήσουμε τι κυβερνήσει. διότι αν πάρει από την Ούνρα μια κυβέρνηση, μια επιστολή, ελπίζω ότι θα επιδείξει περισσότερο πνεύμα ευαισθησία. Αυτό απλώς ήθελα να πω. Ναι, ναι, ναι. Συγγνώμη, συγγνώμη. Ίσως ε, παρανόησα αυτό που είπατε. Ναι, βεβαίως. Ακόμη και αυτό είναι κάτι το οποίο ε, θα μπορούσαμε να κάνουμε να στείλουμε ένα γενικότερο σημείο. αλλά ελπίζουμε ότι η Παλαιστινιακή Αρχή είναι η αρχή για όλους, δεδομένου ότι είναι η Παλαιστινιακή κυβέρνηση και με αυτοί εκπροσωπούν και το ποιολόγια τους Παλαιστινίους. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε να βοηθήσουμε, αλλά είναι κάπως λεπτό το θέμα για μας, διότι πιστεύουμε ότι αυτοί θα πρέπει για το θέμα αυτό να αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Βεβαίως τους υποστηρίζουμε κάνοντας ε, κάτι τέτοιο όπως λέτε εσείς ή αν υπογραμμίσουμε ότι υπάρχει ανάγκη να ενεργήσουμε αυτόν τον τρόπο και στο παρελθόν και φοιτητέ από την Παλαιστίνη και κάποιοι πρόσφυγες πήραν ε, υποτροφίες για να πάνε να σπουδάσουν σε άλλες χώρες και στη ΣΥΠΑ και δεν τους επετράπει να φύγουν. Αυτό είναι κάτι το οποίο το καταδικάσαμε και εκφράσαμε τις αρέσκειά μας δημοσίως προς το Ισραήλ, Φερρυπίν. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει στην ε, συγκεκριμένη περίπτωση για τους φοιτητές να είναι πιο εύκολο να βγουν από την περιοχή αυτή, από την λωρίδα της. Μαζαλά. Ε, προτιμούμε για τους Παλαιστινίους να σύνολό τους να μιλήσει η Παλαιστινική Αρχή, η Παλαιστινική Κυβέρνηση. Τώρα, η γερμανική κυβέρνηση αν έχει κάνει, με ρωτήσατε, συγκεκριμένες προτάσεις. Όπως ξέρετε, ε, είναι δύσκολα τα πράγματα. Η διάσκεψη της Ρώμης έγινε την ημέρα που ορκίστηκε η κυρία Μέρκελ. Αλλά Ξέρουμε ότι υπάρχει υποστήριξη, θέλω να μας ε, βοηθήσει η γερμανική κυβέρνηση όταν αναλάβει επισήμως τα καθήκοντά της. Ήδη υπάρχουν συνεχιζόμενες ομιλίες και για θέματα που αφορούν τον προπολογισμό και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και ένα τράστε το οποίο θα χειρίζεται η Παγκόσμια Τράπεζα και κυρίως για θέματα που αφορούν τους νέους. Πιστεύω ότι θα πρέπει αυτό το κονδύλι, αυτό το τράστα να δημιουργηθεί και να συνεισφέρουν και άλλες χώρες και είναι κάτι το οποίο ε, χαιρετίζουμε, αλλά βεβαίως θα έρθουμε σε επαφή με τη νέα γερμανική κυβέρνηση. Τώρα, όπως ελέγχθη, να έρθουν κάποιοι νέοι μαθητές από τη Γάζα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Ματίας Σμάλε θα πρέπει να το δει αυτό, αλλά βεβαίως ε, οποιαδήποτε σχολείο και στην, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γερμανία, στην ε, Φλάνδρα, ε, γιατί να μην το κάνουμε και αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να το δούμε και θα είναι για μας μία εξαιρετική ευκαιρία και με μεγάλη υπερηφάνεια να το κάνουμε αυτό. διότι θα είναι και μέσω των συζητήσεων που θα γίνουν και για αυτούς η εξαιρετική ευκαιρία που τους προσφέρεται να μάθουν περισσότερα για την ε, Ευρώπη. Θα μας πούνε τι κάνουν και θα μάθουν και από εμά. Μαργαρετ, νομίζω ότι εσύ ανέφερε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο γνωρίζω αλλά δεν θα μπω σε λεπτομέρεια και πάλι σας ευχαριστώ που μας καλέσατε και μας δείτε την δυνατότητα να παρουσιάσουμε το όλο θέμα. Δεν έχει τελειώσει η κρίση, χρειαζόμαστε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ε, ξέρουμε ότι θα αποστελεί επιστολή και στις περαιτέρω συζητήσεις που θα γίνουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ληφθεί αυτό απόψη παρά το γνωστό ότι είναι νωρίς ακόμη για τον προπολογισμό. Ελπίζω λοιπόν ότι θα ε, μπορέσει να υποφεληθεί ενδεχομένως η Ούνρα από κάποια αδιάθετα ποσά, αλλά πρέπει να σας πω ότι δεν μπορούμε ίσως να περιμένουμε πάρα πολύ, διότι πραγματικά μας έχει ε, μας χτυπάει την πόρτα με επιμονή τέλος Ιουνίου η κρίση. Για την παρουσία και την ενημέρωση να πω ότι ε, και από την ενημέρωση που είχαμε από εσά ε, και από τον ε, ε, κύριο Σμέιλ στην Γάζα ε, καταλαβαίνουμε πόσο επίγουσες είναι οι ανάγκε. Ότι είμαστε μπροστά σε μια ανθρωπιστική κρίση, η δουλειά της ΟΥΝΡΑ είναι ε, αναγκαία για εκατομμύρια από ανθρώπους ε, εκεί στην Μέση Ανατολή. Εμεί στράζουμε πέραν από το ψήφισμα ε, που εγκρίναμε τον περασμένο Φεβρουάριο ε, θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας και αναφερθήκε στην επιστολή αλλά και με κάθε ευκαιρία θα τονίζουμε και προς την Επιτροπή και προς το Συμβούλιο και προς κάθε κατεύθυνση ότι χρειάζεται να στηριχθεί η Ούντρα, είναι απαραίτητη για να ε, και για την πορεία ειρηνευσή, αλλά είναι απαραίτητη για να αντιμετωπιστεί άμεσα η ανθρωπιστική κρίση. Ευχαριστούμε και πάλι για την παρουσία σα και για την ενημέρωση. Αγαπητοί συνάδελφοι, η επόμενη συνεδρία μα θα πραγματοποιηθεί στο Στρασβούργο στι 19 Απριλίου από τι 9 μέχρι τι 10.30. Ευχαριστώ όλου για την παρουσία σα σήμερα εδώ και να ευχαριστήσω και του διερμηνεί για τη συμβολή του ώστε να πραγματοποιηθεί η σημερινή μα συνεδρία με όλες τις ομαλές συνθήκες. Ευχαριστώ και πάλι.